Goed, eh, eh, Αντικαθιστώ τον κύριο Τόιβερ σήμερα το πρωί, ο οποίος ε, είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση, κάποια άλλη συνεδρίαση. Αύριο θα είναι εδώ όμω. Καλώς ήρθατε λοιπόν όλοι. Έχετε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης μπροστά σας, φαντάζομαι. Μια παρατήρηση έχω να κάνω μόνο στο σημείο 7 πρέπει να αναβληθεί. Το έχει ζητήσει ο ίδιος εισηγητής, ο κύριο Ριβελίνη, ο οποίος εξακολουθεί να δουλεύει πάνω στην γνωμοδότησή του αυτή. Άρα δεν θα μπορέσουμε να εξετάσουμε σήμερα αυτή την έκθεση. Κατά τα άλλα, συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη. Καλώς. Ανακοινώσει του Προέδρου τώρα, το σημείο 2 δηλαδή. Στο News Brief έχετε τις γλώσσες που έχετε σήμερα. Λέει επίση ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μα και έχουμε και δύο νέα μέλη στην Επιτροπή μας, στην Γραμματεία της Επιτροπής μας. Είναι η κυρία Κάρολα Ενοσάλιβαν η μία και ο κύριο Ολιβιέ Σοτιέρ είναι ο άλλος. Καλώς ήρθατε και οι δύο στην Γραμματεία της Επιτροπή μας. Προσβλέπουμε σε πολύ καλή συνεργασία μαζί σας. Στη συνέχεια πάμε στο σημείο που είναι η έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασής μας, της συνεδρίας δηλαδή η και 18 η Ιουνίου. Ω συνήθω, αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλο τη συνεδρίασή μα, θεωρούνται εγκεκριμένα. Και έτσι περνάμε στο πρώτο ουσιαστικό σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η ειδική έκθεση αριθμός 7 κάθετος 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. το ελεκτικό συνέδριο και ο τέος συναδελφός μας, ο κύριος Ιτάλα, έχουν ετοιμάσει την έκθεση αυτή και συγητής από την Επιτροπή μας είναι ο κύριος Μέλντερ. Να δώσουμε το λόγο Γιάννη στο ελεγκτικό συνέδριο πρώτα. Να ακούσουμε για την ειδική έκθεση και μετά θα πάρει το λόγο η συγητής. Και θα δούμε βέβαια ποιος άλλο θέλει να πάρει το λόγο, μπορεί να γραφτεί στον κατάλογο μιλητό. Παρακαλώ, κύριε Ιτάλα, Καλώ ήρθατε. Έχετε το λόγο εκ μέρου του ελεγκτικού συνεδρίου, λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την ειδική αυτή έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ήδη τώρα ε, είναι, αυτή ε, τη στιγμή είναι πολύ επίκαιρο το θέμα διότι προσπαθούμε να πάρουμε άλλες αποφάσεις οι οποίες θα επανέλθω αργότερα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Συστάθηκε το 2006 για να καταδείξει αλληλεγγύη προς τους εργαζόμενους που απολύονται και ο στόχος είναι να διευκολύνει την επανένταξη στην απασχόληση με τον εργαζομένο αυτόν με την παροχή κάποιων συνεισφορών, ε, κάποιων δεσμών για και εδώ περιλαμβάνονται μέτρα για την αγορά εργασίας, κατάρτιση, ενίσχυση αυτοπασχόληση κτλ. Επίσης πολλές φορές περιλαμβάνουν στήριξη του εισοδήματος και η πρώτη εφαρμογή ε, για το ταμείο αυτό έγινε το 2007 από τη Ρενό και εμείς Πήγαμε σε τέσσερα κράτη-μέλη σαν ελεγκτικό συνέδριο και ελέγξαμε την κατάσταση στα τέσσερα κράτη-μέλη στα οποία χρησιμοποιήθηκε και άλλες τέσσερις χώρες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει γιατί άλλες χώρες δεν έχουν χρησιμοποιήσει το ταμείο καθόλου. Πριν να σας αναφέρω αποτελέσματα, να τονίσω κάτι τι. Ο στόχος, το ταμείο αυτό και η στόχοι του είναι γενικά αποδεκτή γιατί έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τους απολυμμένους εργαζόμενους να ενταχθούν και πάλι στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα να αναφέρω τέσσερα πράγματα. Να πω ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία όπως παραδείγματο χάνει ότι εδώ καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι και αλλά δεν είναι, υπάρχουν και αρνητικά σημεία Παραδείγματο χάρη χρειάζονται στοιχεία όμως τα οποία, δεν, τα οποία δεν μας δίνονται για να αξιολογήσουμε την κατάσταση από τις 8 χώρες που ε, επισκεφτήκαμε προσπαθήσαμε να εξάγουμε μετρήσιμα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους. Η... Το Ταμείο υποστηρίζει πολλά και χρήσιμη, την εφαρμογή πολλών και χρήσιμων μέτρων αλλά επίσης πάρα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν από τα κράτη-μέλη. Από τις 89 περιπτώσεις τις οποίες ελέγξαμε ένα τρίτο των κονδυλίων πήγαν σε στήριξη του εισοδήματο. Σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από το 50% πήγαν για τέτοιου είδους μέτρα τα μέτρα κατάρτισης που κατά τη δική μου προσωπική άποψη θα έπρεπε να είναι τα πιο σημαντικά μέτρα που χρηματοδοτούνται ε, τα μέτρα κατάρτισης λοιπόν ε, πήραν πολύ λίγα χρήματα η ενδιάμεση αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μόνο 26% των δαπανών του Ταμείου πήγαν στην κατάρτιση και εδώ αξίζει να πούμε ότι όλα τα μέτρα του κανονισμού του Ταμείου μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι σημαντικό επίσης να σημειώσουμε ότι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει αμέσ, άμεσα ορισμένα προβλήματα αλλά οι διαδικασίες καθυστερούν ο μέσος όρος είναι 41 εβδομάδες για την ε, παροχή της πραγματικής ε, βοήθειας και αρκετά κράτη-μέλη ακριβώς γι' αυτό το λόγο είπαν ότι δεν έκαναν αιτή στο Ταμείο καθόλου. Κύριε Πρόεδρε, Βάσει των πορισμάτων του ελεκτικού συνεδρίου κάνουμε τις εξής συστάσεις. Πρώτον, τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχουν στοιχεία ενημερωμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τα, το κατά πόσο να πετεύθησαν οι στόχοι και να μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των διαφόρων μέτρων. Ο νομοθέτης θα πρέπει ίσως να περιορίσει τη χρηματοδότηση για εκείνα τα μέτρα τα οποία προσφέρουν πρόσθετη αξία αν θέλετε, ευρωπαϊκή αξία άλλο και όχι κατά πλειοψηφία σε στήριξη του εισοδήματος υπάρχουν, μπορεί να ίσως να πρέπει να οριστεί και κάποιο όριο εδώ. Τέλος, οι νομοθέτες, ο νομοθέτης θα πρέπει να σκεφτούν ότι υπάρχει εναλλακτική λύση, σαν εναλλακτική λύση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, για να βοηθηθούν αυτοί οι οποίοι απολύονται μαζικά. Ξέρουμε ότι η μεγάλη απόφαση ήδη έχει πάρθει για τη συνέχιση του Ταμείου. Όμως θα πιστεύουμε ότι θα πρέπει οι συστάσεις που κάνουμε θα πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη και ιδιαίτερα όταν θα γίνει η διάμεση έκθεση για το επόμενο πρόγραμμα, για το επόμενο χρονικό πλαίσιο. Κύριε Πρόεδρε, η ειδική αυτή έκθεση και το πότε γίνεται η έκθεση αυτή ε, πρέπει να λάβει ε, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Πρέπει να είναι μια χρονική στιγμή που υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να παρθούν ορισμένες αποφάσεις και από τον νομοθέτη κτλ. Για τούτη εδώ την ειδική έκθεση να σας πω ότι κανονικά θα έπρεπε η έκθεση αυτή να δημοσιεύει θα έπρεπε να δημοσιευθεί αρχές του 2014 ε, γιατί θα είχαμε περισσότερα στοιχεία ίσως τότε για να, στα οποία να βασιστούμε ήταν λοιπόν ατυχές το γεγονός ότι έγινε τώρα ο έλεγχος για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε λοιπόν σωστά για τις τελικές διαπραγματεύσεις για το νέο ταμείο αναγκαστήκαμε να επιταχύνουμε τις εργασίες μας και χάρη των συνεργατών μου και των, της ομάδας του ελεκτικού συνεδρίου πήγαν καλά τα πράγματα πρέπει να τους ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω επίσης και την Κομισιόν γιατί χωρίς τη βοήθεια της Κομισιόν δεν θα συστούσαμε την ειδική έκθεση σήμερα. Παρόλο λοιπόν που η έκθεση αυτή ίσως ε, έρχεται καθυστερημένη για τη συζήτηση του πολιετούς προγράμματος ε, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η έκθεση αυτή έγινε έξι μήνες νωρίτερα από ό,τι θα γινόταν κανονικά και ε, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν να την κρίνουμε. Κλείνοντας την παρουσίασή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε τον κύριο Μίλντερ για τη συνδρομή του όπως και παλιότερα ε, είχαμε πολύ καλή συνεργασία και το έγγραφο εργασίας που ετοίμασε και εκείνο είναι καλή βάση για τις μελλοντικέ σας εργασίες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο πρώτα στον εισηγητή. Ο κύριος Ζούμπη έχει ζητήσει άλλος, ο κύριος Σέπινγκ, άλλος. Όχι, καλώς. Ο εισηγητή λοιπόν πρώτα και μετά οι δύο συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Α, και εσεί. Και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, Γιάν Μέλντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο, ιδιαίτερα δε τον κύριο Ιτάλα, για την ε, καλή δουλειά αλλά και την καλή συνεργασία που είχαμε. Νομίζω ότι ε, το αποτέλεσμα ε, είναι σωστό, οι γενικές, τα γενικά συγγνώμη συμπεράσματα είναι όρθα και τα συμμερίζομαι. Βεβαίως υπάρχουν πάντα στοιχεία τα οποία μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω. Πρώτα απ' όλα ο στόχος του Ταμείου είναι να βοηθήσει τους απολυμμένους εργαζόμενους, να τους καθοδηγήσει σωστά, έτσι ώστε να μπορέσουν να επανατοποθετηθούν στην αγορά εργασίας. Ε, ε, οτιδήποτε και αν σκέφτεται κανείς για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, σε ένα νέο ε, πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα, αυτά έχουν ήδη αποφασιστεί και επομένως τα δύο αυτά ταμεία για τα οποία γίνεται γίνεται λόγος, θα πρέπει να ε, έχει αποφασιστεί ότι θα πρέπει να συνεχίσουν ε, την δράση τους. Αλλά ε, ο βαθμός χρηματοδότησης να είναι 50 με 60% στο, για το Ταμείο Προσαρμογής και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να φτάνει μέχρι το 85%. Εξηγούμε. Ε, υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αποσαφινιστούν στον τριμερή διάλογο ε, που λαμβάνει ε, χώρα υπό την αιγίδα μιας άλλης κοινοβουλευτικής επιτροπής μαζί βεβαίως με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Θα πρέπει στη διάρκεια αυτού του τριμερούς διαλόγου να προσέξουμε έτσι ώστε τα γενικά συμπεράσματα ε, του ελεγκτικού ε, συνεδρίου να ληφθούν υπόψη και συμφωνώ με το ελεγκτικό συνέδριο που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή ποσοστοποίηση και αποσαφήνιση των στόχων. Θα πρέπει κανείς να ξέρει ε, σε τι αποσκοπεί και τι θέλει να επιτύχει. Αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω και θα πρέπει να υπογραμμιστεί περισσότερο. Ότι δηλαδή το Ταμείο ε, Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι συμπληρωματικά. Επίση, ότι θα πρέπει ε, η ε, διαφορά μεταξύ των οποίων όσον αφορά συγκεκριμένα στοιχεία θα πρέπει να προγραμμιστεί περαιτέρω. 41 εβδομάδες είναι το χρονικό όριο. Είναι πάρα πολύ μακρύ κατά την άποψή μας. Είναι ένας χρόνος σχεδόν. 10 μήνες, σε πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά μέχρι τότε νομίζω ότι τα πράγματα έχουν, στους 10 μήνες δηλαδή αυτούς που μεσολαβούν, τα πράγματα μπορεί να έχουν πάει πάρα πολύ άσχημα. Ε, επίσης, εξωτερική χρηματοδότηση, ένα τρίτο του ταμείου χρησιμοποιείται για την αποζημίωση ε, των ε, μισθών. Αναρωτιέμαι, είναι καλός τρόπος να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα. Επίσης, Έχω και κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Οι 41 εβδομάδες. Καλό θα ήταν ε, να υπάρξει στον επόμενο κανονισμό ε, μία άλλη προθεσμία. Δηλαδή να πούμε αν σε δύο-τρεις μήνες δεν μπορεί να γίνει τίποτα τότε να το ξεχάσουμε. Γιατί αυτός είναι ε, ένας λογικός χρόνος, ένα λογικό χρονικό διάστημα, οι δύο-τρεις μήνες έτσι ώστε να αποφασίσει η Κομισιόν τι μπορεί να γίνει. Έχω την ε, εντύπωση κύριε Πρόεδρε και, και ζητάω και βλέπω τις συστάσεις που έχω υποβάλει. Νομίζω ότι αναφέρθηκα στις ε, προτάσεις που κάνω. Να πω ότι σε γενικές γραμμές ε, τεκμέρεται θετική η θέση του Συμβουλίου και η στάση ελπίζουμε ότι στην επόμενη αξιολόγηση ε, θα είναι πολύ σημαντική η θέση του ελεγκτικού συνεδρίου. κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Ιτάλα και τον κύριο Μιλντερ για την εισαγωγή που μας έκαναν στο θέμα αυτό του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που είναι πάρα πολύ σημαντικό ιδιαίτερα εν ώψη υπό το φως μάλλον της ενεργείας των ε, νέων. Η Siemens παραδείγματο χάρη θέλει να απολύσει 10.000 άτομα, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πρόκειται να απολυθούν και όχι μόνο από τη Siemens. Ε, είναι πολύ σημαντικό και για τους άνεργους και για αυτούς που πρόκειται να απολυθούν στο μέλλον να τους δώσουμε εναλλακτικέ λύσεις, κατάρτισης, επιμόρφωσης, διαβίου μάθης κτλ. Αν κατάλαβα καλά γύρω στο 25% των κονδυλίων του Ταμείου δόθηκε για εκπαίδευση. Ερώτηση, τι, πόσο αποτελεσματικά ήταν τα κονδύλια αυτά, ήταν καλής ποιότητας η κατάρτιση, βρήκαν δουλειά στο τέλος οι άνθρωποι που την παρακολουθούν ακολούθησαν. Μήπως υπάρχει στην Ευρώπη ένα σύστημα best practice ή ένα σύστημα benchmark βάσει του οποίου μπορούμε να κρίνουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή για να δούμε ίσως πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα στο μέλλον. Και προβλέπετε... Ε, προβλέπετε να γίνει κάτι τέτοιο και θα ήθελα κατάλαβα ότι ο μέσος όρος είναι 41 εβδομάδες ε, θα ήθελα να μου πείτε όμως ποια ήταν η πιο γρήγορη διαδικασία και θυμάστε και την οδηγία για τις απληρωμές ε, που έχει τις 90 μέρες έτσι δεν ξέρω αν συνδέονται αυτά Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Έπινγκ Ευχαριστώ πρόεδρε Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ το Ελεκτικό Συνέδριο για την έκθεσή του. Πάντα με ενδιαφέρουν δικές εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, διότι υπογραμμίζουν πράγματα τα οποία συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραβλέπουν. Το Ταμείο λοιπόν για την παγκοσμιοποίηση είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε πάντα με σκεπτικισμό. Είμαστε κατά σε κάθε πρόταση πληρωμών που έρχονται από το Ταμείο. Και τώρα με αυτά που λέει το ελεκτικό συνέδριο επιβεβαιώνομαι. Η κυρία Ματέρα, η εισηγήτρια μέχρι τώρα πάντα υποστήριζε τις ε, εκθέσεις και τώρα θεωρούμε ότι είναι το Ταμείο αυτό κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί από, να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις. Φυσικά οι προθέσεις είναι καλές, είναι θετικές, είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν την δουλειά τους. Από την έρευνα όμως που γίνεται βλέπουμε ότι ο στόχος δεν είναι τόσο ξεκάθαρος. Δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία που θα θέλαμε και όπως περιμένουμε ένα μεγάλο μέρος χρησιμοποιείται για τη στήριξη του εισοδήματος και ένα μικρό μέρος μόνο για την κατάρτιση, την ε, επανακατάρτιση των ανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ισχνό, κάτι το οποίο φοβόμασταν και γι' αυτό ακριβώς και δεν το θέλαμε. Συνεπώ, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι έχει αποτύχει το Ταμείο αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πιστεύει ότι με μικροδιαχείριση μπορεί από τις Βρυξέλλες να κατευθύνει το τι γίνεται στις επιχειρήσεις και ότι το ταμείο αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε να συμπεριληφθεί στο κοινωνικό ταμείο και να μην έχουμε δύο διαφορετικά ταμεία. Δεν μας χρειάζεται ένα ξεχωριστό ταμείο, το οποίο δημιούργησε ίσως πολλές προσδοκίες, αλλά τελικά δεν έχει πετύχει αυτά τα οποία θέλαμε. Είναι πια γεγονός. Καλό είναι λοιπόν να παραιτηθούμε από αυτό το ταμείο. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος. Ε, η κυρία και έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τον εισηγητή μας για την ειδική αυτή έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την παγκοσμιοποίηση. Πολλές ε, εκθέσεις αναφέρουν διάφορα ενθαρρυντικά για το Ταμείο αυτό. Συγχρόνω όμως πρέπει να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο, να το απλοποιήσουμε και να είμαστε πιο επικεντρωμένοι σε συγκεκριμένους στόχους. Το Ταμείο αυτό περιγράφεται ως ένα εργαλείο το οποίο παίρνει πάρα πολύ χρόνο να εγκρίνει κονδύλια, εφαρμόζει τα μέτρα πολύ αργά, δεν διέπεται από ευελιξία, υπάρχει και το ποσοστό της συγχρηματοδότησης που είναι χαμηλότερο από το κοινωνικό ταμείο, μιλάει για προχρηματοδότηση η οποία όμως δεν έχει εισαχθεί όπως πρέπει κλπ. Συνεπώς, όταν διαβάζουμε όλη αυτή την περιγραφή, δεν μπορούμε να συνδέσουμε την περιγραφή αυτή με τα αποτελέσματα που θέλουμε να είναι άμεσα από το Ευρωπαϊκό αυτό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Γι' αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά παρετέρω και να δούμε τι αλλαγές πρέπει να επιφέρουμε σε αυτό, ώστε πιο στοχευμένα να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση. Έπειτα αν δούμε το τι έχει τελικά χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο αυτό και από το Κοινωνικό Ταμείο, διαπιστώνουμε ότι τα ίδια πράγματα χρηματοδοτούνται. Ότι δηλαδή γενικά αρρωγή στην απασχόληση, κατάρτιση, στήριξη για την επιχειρηματικότητα, επιδοτήσεις κτλ. Είναι πράγματα τα οποία χρηματοδοτούνται και από τα δύο ταμεία. Καλό είναι να δούμε ποιο από τα δύο ταμεία έχει τα καλύτερα αποτελέσματα και το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση είναι επικεντρωθεί σε δύο-τρεις μόνο στόχους, εκεί όπου μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό. Ίσως τότε το Ταμείο αυτό να μπορέσει να δράσει πιο γρήγορα και να μην καθυστερεί. Επίσης το θέμα της απλοποίησης είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως θα μπορούσαμε την έγκριση αυτή να την κάνουμε βάση του περιεχομένου. Δηλαδή να είναι κάποια light διαδικασία, μετά από την οποία να μπορεί να ξεκινήσει η εφαρμογή και μετά να ξεκινάει η ενδελεχής διαδικασία έγκρισης. Γιατί αν χρειάζονται 30 εβδομάδες, 8 μήνες δηλαδή, φαντάζεστε, είναι ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό στο κάτω-κάτω μέσα σε 30 εβδομάδες μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες στην αγορά. Οπότε τα προτινόμενα μέτρα να μην είναι πια τόσο αποτελεσματικά αν τεθούν σε εφαρμογή 30 ή ακόμα περισσότερους μήνες αργότερα από τη στιγμή που προτείνονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς, παρακαλώ. Όχι. Ωραία. Ακούσαμε λοιπόν διάφορες απόψεις που πάνε από το να το καταργήσουμε το Ταμείο μέχρι να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε τις διαδικασίες έγκρισης. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως θέλει να αντιδράσει. Α, ναι. Ποιος, παρακαλώ. Παρακαλώ, πείτε ποιος είστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Τετλαφάκα και είμαι υπεύθυνο διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση για το Ταμείο αυτό. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για το εξαίρετο έργο του. Όπως είπε το ελεγκτικό συνέδριο εξάλλου, εκπονήθηκε η έκθεση αυτή μέσα σε πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας. Εξάλλου είναι και προς το δικό μας το συμφέρον να έχουμε μια καλή και στέρεα ανάλυση του Ταμείου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου και ποσοτικά αλλά και όσον αφορά την ανάλυση μπορούμε να συμφωνήσουμε και συμφωνήσαμε να δεχτούμε τα περισσότερα από τα σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου. Βέβαια πρέπει να δούμε το ταμείο αυτό μέσα σε κάποια προοπτική για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα αρνητικά σχόλια που έγιναν. Βλέπετε, είναι ένα από τα μέτρα το οποίο δεν εμπίπτει μέσα στις πολυδιανομιστικές ε, προοπτικές κατευθείαν με τη στενή έννοια του όρου, αλλά γενικότερα στον προπολογισμό. Οπότε τα μέτρα είναι στοχευμένα. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου δείχνει ποια είναι τα μέτρα εκείνα τα οποία βοήθησαν τον κόσμο που επλήγει από απολύσεις. Αναφέρεται επίσης στην έκθεση αυτή του Ελεκτικού Συνεδρίου ότι υπήρξε ε, συντονισμός ανάμεσα στις δράσεις του Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση και του Κοινωνικού Ταμείου, κάτι το οποίο ήταν θετικό. Κάποιες χώρες προτιμούν το Κοινωνικό Ταμείο, κάποιες άλλες προτιμούν το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Αναγνωρίζει επίσης το Ελεκτικό Συνέδριο ότι χώρες μέλη μάλλον ικανοποιημένες δηλώνουν από τη στήριξη που είχαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος δεν υπήρξαν θέματα ε, νομικά τέτοιες δυσκολίες όσον αφορά την επιλεξιμότητα των ε, μέτρων. Τώρα οι συστάσεις που γίνονται έχουν να κάνουν με τη διαθεσιμότητα των ε, στοιχείων μεταξύ άλλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί και γι' αυτό έχει ήδη στη νέα μας πρόταση συμπεριλάβει κάποιες διατάξεις ώστε στον τριμερή διάλογο να μπορούμε να δώσουμε τα στοιχεία αυτά. Η διαθεσιμότητα των στοιχείων, βλέπετε, έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τις χώρες μέλη. Προχωρώντας, θα διαπιστώσουμε ότι ηλεκτρονικά όλο και περισσότερα στοιχεία θα μπορούμε να έχουμε. Αρχίσαμε λοιπόν τη διαδικασία εφαρμογής, αναβαθμίζοντας και εξυγχρονίζοντας τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού συστήματος, κάτι το οποίο θα βοηθήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε τα στοιχεία που ζητάμε. Απευθεία σχεδόν. Φροντίσαμε και για προπολογισμό όσον αφορά την τεχνική αρρωγή για την αναφορά στοιχείο. Και στον νέο κανονισμό γίνεται η σύσταση. Όλα αυτά συζητήθηκαν στον άτυπο τριμερή διάλογο. Η έκθεση πάντως του Λεκτικού Συνεδρίου να ξέρετε ότι μας βοηθάει στις συζητήσεις που έχουμε με τους δύο συνομοθέτες. Όσον αφορά τώρα το θέμα της περιορισμένης προστιθέμενης αξίας, η επιτυχία που έχουμε σε κάποιους τομείς δείχνει ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα των μέτρων. Είπατε, μα δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Μα έχουμε ετοιμάσει έκθεση για το 2012 που δείχνει ότι το 50% των καταρτιζόμενων βρήκαν τελικά δουλειά παρά την κρίση. Ε, πολύ θα θέλαμε να είχαμε καλύτερο ακόμα αποτέλεσμα και πιστεύω ότι όταν βελτιωθεί κάπως το οικονομικό κλίμα, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Πάντως και εμείς προτείνουμε στόχους στο νέο κανονισμό όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργαζομένων. Τώρα το ελεκτικό συνέδριο επίσης υπογραμμίζει πολύ ένα πολύ σημαντικό θέμα που και εμείς το αναφέρουμε στις προτάσεις μας για τον νέο κανονισμό όσον αφορά τις παροχές για το 50%. Τώρα θα μου πείτε γιατί 50% ενώ είχαμε 30% κατά μεσόρο. Πιστεύουμε ότι δεν θα είναι μεγάλο πρόβλημα κάποιες περιπτώσεις είναι πάνω από 50% και τότε υπάρχει ανισορροπία. Γιατί είναι 30% αυτό που θα μπορούσαμε να δεχθούμε, γιατί είναι όλα που έχουν να κάνουν με τις επιδοτήσεις εισοδήματος και με την επανακατάρτιση. Δεν πληρώνουμε δηλαδή τους ανθρώπους για να μην κάνουν τίποτα, για να κάθονται. Αυτή η εντύπωση δεν είναι ορθή. Όταν καταρτίζονται όταν ε, αναλαμβάνουν ε, κάποια νέα, ε, ξεκινάνε καινούργια μαθήματα, ή κάποιο είδους κατάρτιση τέλος πάντων, τότε έχουν τις επιδοτήσεις αυτές τις εισοδηματικές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τώρα σε τι βαθμό αυτό αποτελεί επικάλυψη με άλλα μέτρα εθνικού χαρακτήρα. Εδώ πρέπει όντως να πετύχουμε μια καλή ισορροπία γιατί δεν θέλουμε να εμποδίζουμε τα κράτη-μέλη, να τους θερήσουμε δηλαδή την ελευθερία που έχουν να διαχειρίζονται όσο γίνεται καλύτερα τα δικά τους μέτρα. Η συζήτηση λοιπόν σε σχέση με αυτήν την επιδότηση του εισοδήματος είναι περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα. Επί της ουσίας συμφωνούμε και εμείς ότι δεν θα έπρεπε να είναι πάνω από 50%. Δεν θα πρέπει να είναι δηλαδή το κύριο στοιχείο του προγράμματος. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό και η σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου μας βοηθάει πολύ και τις δίνουμε βάση. Όσον αφορά τώρα το ταμείο, τη σχέση μάλλον του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης με το Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επ' αυτού αναφέρθηκε και ακούστηκαν διάφορα επιχειρήματα οι επακεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισαν. Εδώ υπήρχε το γιατί 50 και 65% η Κομισιόν 85% εξαρτάται από τα κράτη-μέλη στο κοινωνικό ταμείο. Μα εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές λογικές παρέμβασης. Και το άλλο είναι ότι είναι δύο διαφορετικοί προπολογισμοί. Έχουμε την συγχρηματοδότηση των εθνικών, ε, ε, της εθνικής αρρωγής και εδώ παρεμβαίνει και το Ταμείο Συνοχής. Η παρέμβαση δηλαδή εδώ είναι εντελώ διαφορετική. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως είπαν κάποιοι, παρεμβαίνει ad hoc, επιπλέον Αν μιλούσε εδώ ως κράτος μέλος και είχα την επιλογή 85% κοινωνικό ταμείο ή 65% ταμείο παγκοσμιοποίησης, θα προτιμούσα τις παγκοσμιοποίησεις, γιατί είναι επιπλέον χρήματα. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει ντοκτορά στην οικονομία για να καταλάβει ότι έτσι υποφελείται. Το πρόβλημα βέβαια μερικές φορές που έχετε είναι ότι η διοικητική ικανότητα των κρατών μελών είναι τέτοια που δυσκολεύεται να διαχειριστεί δύο διαφορετικά προγράμματα. Είναι γεγονός. Για το χρονοδιάγραμμα και τις 41 εβδομάδες που είναι ο μέσος όρος. Να σας εξηγήσω λιγάκι τι κρύβεται εδώ από πίσω. Για κάθε περίπτωση, γιατί δεν είναι προκαθορισμένος ο προϋπολογισμός, πρέπει κάθε φορά να λαμβάνεται απόφαση από τους συνομοθέτες. Πάντως έτσι ήδη εισαγάγεται η μακρά αυτή περίοδος. Γι' αυτό και καθυστερεί πολλές φορές. Στη συνέχεια τα κράτη-μέλη μπορούν να αρχίσουν να χρηματοδοτούν ένα μέτρο ακόμα και πριν να έχει κάνει την πρόταση κομισιόν και πριν οι αρχές επί του προπολογισμού να έχουν πάρει την απόφασή τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την συγχρηματοδότηση για να αρχίσουν να χρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Η μακρά περίοδος δεν εμποδίζει τους εργαζόμενους να υποφεληθούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα που πρέπει να περάσει εδώ. Πάντως οι 41 εβδομάδες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Πράγματι, στηρίζουμε το Κοινοβούλιο στον τριμερή διάλογο που θέλει σαφείς προθεσμίες. Θέλουμε και εμείς να μειωθούν οι 41 εβδομάδες κατά μέσο όρο. Κατά 10 εβδομάδες, για να σας δώσω μια ιδέα του τι είναι εφικτό. Αν γίνει αυτό θα είναι μεγάλο βήμα. Και προσπαθούμε επίσης αυτή την εποχή να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Μερικές φορές η μακρά περίοδος οφείλεται και στο γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν όλες τις πληροφορίες. Συνεπώς εδώ πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη, δεν δίνουν μάλλον τα κράτη-μέλη τις πληροφορίες όλες που χρειαζόμαστε. Πρέπει λοιπόν να τα πιέσουμε να μας δίνουν πιο γρήγορα τις πληροφορίες τους. Να τις έχουμε όλες, να μην χρειάζεται να τις ζητάμε ξανά και ξανά, έγκαιρα. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα στοιχεία της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου, όπως επίσης και τα περισσότερα σχόλια που ακούστηκαν εδώ στην αίθουσα από τους ευρωβουλευτές. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση εξυπηρετεί έναν πολύ σημαντικό σκοπό. Είναι μια πράξη αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για σημαντικές περιπτώσεις απολύσεων, ποιοι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Γιατί λέτε δεν μπορούμε να έχουμε ένα άγγερο σύστημα συναγερμού προειδοποίησης. Είναι κάποιες χώρες που μπορούν και μπορούν να αρχίσουν να δουλεύουν χρησιμοποιώντας το κοινωνικό ταμείο πριν το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. φροντίζουν έτσι για την απασχολησιμότητα. Αλλά είναι γεγονό ότι δεν χρειάζεται να περιμένουν οι χώρες να χάσει τη δουλειά του κάποιο για να παρέμβουν. Φτάνει να υπάρχει απόφαση που λέει ότι για παράδειγμα θα κλείσει μια επιχείρηση, ότι δηλαδή θα χάσει τη δουλειά του ο εργαζόμενος. Άπαξ και γίνει γνωστή η απόφαση αυτή, τότε αμέσω μπορεί να μπει η διαδικασία στο αυλάκι. Κατά τα άλλα, ετοιμάζουμε η Επιτροπή δηλαδή μια έκθεση για την ε, ποιότητα της πολιτικής προσαρμογής. Είναι κάτι που θα προχωρήσει στα πλαίσια της έκθεσης ΕΡΚΑΣ. Ξέρω ότι μακρηγόρησα, αλλά αισθάνθηκα ότι έπρεπε να μπω στις τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί μερικές φορές είναι σημαντικές για να καταλάβει κανείς και να σχηματίσει ολόκληρη την εικόνα. Πάντως η συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο ήταν ειλικρινά πάρα πολύ χρήσιμη για μας. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Νομίζω ότι τους ε, εκπροσωπώ εδώ, ε, άμα πω, ότι ήταν ιδιαίτερα επεξηγηματικά τα σχόλιά σας και οι παρατηρήσεις σας και σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας άλλος εδώ που θέλει το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Οπότε θα δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Ιτάλα να αντιδράσει και μετά στον εισηγητή για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις ε, που υποβάλλετε. Νομίζω ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον εισηγητή και αυτό είναι κακό. Καλό, συγγνώμη να πω για μία ακόμα φορά ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε στο ποιο, ποια μέτρα ήταν τα καλύτερα, γιατί δεν υπήρχαν τα απαραίτητα συγκρίσιμα στοιχεία και όλα τα εργαλεία πληροφόρησης. Εκατό περίπου ε, απολυμμένοι ε, στα πλαίσια μαζικών απολύσεων ε, μπόρεσαν να ε, χρηματοδοτηθούν. Only the figure. Και επίσης όσον αφορά τα χρήματα, 26% του Ταμείου Προσαρμογής ε, στην Παγκοσμιοποίηση καταναλώθηκε, χρησιμοποιήθηκε ε, για προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές. Εδώ βλέπετε τα στοιχεία. Έχουμε στο σημείο 14 τα στοιχεία. Ε, το, καλύτερο, το, το, καλύτερο αποτέλεσμα το είχε η Λιθουανία με 59%. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τέλος ο Γιάννη Μέλντερ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι πολύ σύντομος. Από ό,τι καταλαβαίνουμε ε, υπάρχει συνένεση ε, κατά το μάλλον τον όσον αφορά τα συμπεράσματα. Είπαμε και προηγουμένως έχουμε τον τριμερή διάλογο υπό την αιγίδα της ε, Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι και η έκθεση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων έτσι ώστε ε, να συμπεριληφθεί ε, κατά κάποιο τρόπο στην διαπραγμάτευση στα πλαίσια του ημερούς διαλόγου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στο σημείο 4 της ημερησίας διατάξεως μπορούμε να... Μάλλον το ολοκληρώσαμε και περνάμε στο 5. Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό Έτος 2014, όλα τα τμήματα. Η συγητής είναι ο Γένς Γκάιερ. Γένς, έχεις γνωμοδότηση, μπορείς να την παρουσιάσεις. Ευχαριστώ πολύ, Μπάρτ. Θα είμαι σύντομος, αγαπητοί Συνάδελφοι, τη διαδικασία τη γνωρίζετε, τη διαδικασία που εφαρμόζουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Σε... Ο εισηγητής για την απαλλαγή σε συνεργασία με την Επιτροπή να ε, αναλαμβάνει την ευθύνη να βάλει τον ε, προπολογισμό για την επόμενη χρονιά. Ε, Προσπάθησε στην στο εγγραφό μου να βάλω όλα τα στοιχεία τα οποία προήλθαν από τη διαδικασία απαλλαγής ε, βασίστηκα σε αυτά τα στοιχεία βασίστηκα επίσης και σε στοιχεία για τα οποία υπάρχει γενικό συνένεση εδώ στην Επιτροπή δηλαδή ενίσχυση των ελέγχων των μηχανισμών ελέγχου να φροντίσουν ε, λέμε βασίσκα στο γεγονό ότι όλοι πιστεύουμε ότι η ευθύνη των κρατών μελών για την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους ε, βιώνουμε ήδη αυτή τη στιγμή την κατάσταση όπου το Συμβούλιο και η Κομισιόν παίζουν ένα είδος πινκ-πονγκ. Το Συμβούλιο ε, ε, κάνει τα σχόλιά του, τα, το ελεκτικό συνέδριο έχει κάνει κάποιες παρατηρήσεις επίσης σχόλια και αρνητικά και όταν τα κράτη-μέλη λένε ότι τελικά η διαχείριση του προπολογισμού ε, δεν είναι καθαρή, δεν είναι αυτή που πρέπει, ε, πραγματικά αναρωτιόμαστε ε, τι κάνουμε. Σε μερικές εβδομάδες θα πάρουμε το έγγραφο από πλευράς κομισιών έγγραφο της Κομισιόν βασίζει το δικό μα το ψήφισμα για την απαλλαγή του περασμένου Απριλίου ένα έγγραφο το οποίο έχει ενοποιημένα στοιχεία από πολλές χρονιές. Ελπίζουμε τα στοιχεία αυτά, τα νούμερα αυτά που θα υπάρχουν εκεί να είναι ε, ε, σημαντικά να δούμε, ελπίζουμε να δούμε πού, ποια λάθη διορθώθηκαν, ποιοι ε, πώς διορθώθηκαν και τι έχουν να πούν τα κράτη-μέλη σχετικά με αυτά. Είναι, τα νούμερα λένε πολλά. Αν θυμάστε πέρσι τι έγινε με την απαλλαγή, ε, τα κράτη-μέλη τι έκαναν πέρσι, το Ηνωμένο Βασίλειο πώς έδρωσε. Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αυτή τη στιγμή να να επιστρέψει 60 εκατομμύρια από κακή διαχείριση των αγροτικών δαπανών. Λοιπόν, συγγνώμη, ε, καταλαβαίνετε τι γίνεται και τα κόμματα στη Γερμανία ε, έχουν, ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν γίνει λάθη Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να τριγυρνάμε και να επικρίνουμε άλλους τον εμείς οι ίδιοι στους δικούς μας τους λογαριασμούς δεν είμαστε εντάξει. Δεν μπορούν λοιπόν κάποια κράτη-μέλη να κατακρίνουν και να επικρίνουν άλλους όταν οι, τα ίδια έχουν να κρύψουν ή, ή ακόμη και αν δεν έχουν να κρύψουν έχουν κάνει λάθη ή δεν κάνουν σωστά τους ελέγχους. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το τονίσουμε αυτό. Αυτή είναι η δουλειά μας. Θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια ποσά λοιπόν με το Συμβούλιο, θα πρέπει να δούμε τι έγιναν με τις ανακτήσεις, να ζητήσουμε κάποια χρήματα από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο βεβαίω θα πει όχι, αλλά βιώνουμε μια οικονομική κρίση, όλοι τη ζουν την κρίση αυτή και από εκεί και πέρα βεβαίω είναι δική μας δουλειά να ενημερώσουμε τον ψηφοφόρο, την ψηφοφόρο για το τι γίνεται με τα χρήματα των φορολογουμένων στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκρέσλ. Έχει ζητήσει το λόγο. Ποιος άλλος. Αντρίασεν. Ποιος άλλος. Και εσείς. Καλώς. Παρακαλώ κύριε Γκρέσλ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει και κάτι τι άλλο που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Εδώ και δέκα χρόνια η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα τρία κράτη-μέλη είναι μονίμως επί δέκα χρόνια στις πρώτες θέσεις αυτών που κάνουν τα λάθη κατάλαβα αυτό που είπε ο συνάδελφος για το Ενωμένο Βασίλειο. Είναι ένα είδος ε, ηρωνίας αυτό. Αλλά εγώ πραγματικά θα ήθελα να μάθω πώς ανέχεται επί δέκα χρόνια η Κομισιόν αυτή την κατάσταση. Τρία κράτη μέλη να είναι μονίμως πρωταθλητές λαθών. Κύριος Αντρέασεν. Η Ευχαριστώ. Θέλω εδώ πέρα να πω σε όλους ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη χώρα που ζητάει μίεση στον κοινοτικό προπολογισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, αν μειωθεί ο προπολογισμό, θα υπάρχουν και λιγότερε πιθανότητε για κατάχρηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι ρόλο παίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχοντας την χρήση των κονδυλίων των ταμείων αυτών, διότι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι τα χρήματα αυτά τα βάζουν στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι στα χέρια των χωρών μελών. Οπότε είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμα και αν τα κονδύλια τα διαχειρίζονται, τέλος πάντων τα προγράμματα εφαρμόζονται στις χώρες μέλη, είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διασφαλίσει πριν δώσει τα χρήματα, πριν ελευθερώσει τα κονδύλια αυτά, ότι τα χρήματα αυτά θα φτάσουν στον σωστό προορισμό τους. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό όμως δεν γίνεται. Και φοβάμαι ότι εξακολουθεί να αποτελεί πηγή των περίφημων σφαλμάτων, τα οποία αναφέρει ξανά και ξανά το ελεγκτικό συνέδριο. Θέλω να αναφερθώ εδώ σε μία πρόταση που γίνεται στην έκθεση Γκάιερ, ο οποίος σημειώνει με ικανοποίηση ότι η σημερινή χρήση 4,5 δις το 2012 είναι. Η διόρθωση αυτή έχει να κάνει με σφάλματα πόσων ετών. Γιατί το ποσό μπορεί να ακούγεται ικανοποιητικό, αλλά αν έχει να κάνει με σφάλματα τα οποία έχουν λάβει η χώρα την τελευταία δεκαετία, ε, δεν θα έλεγα εγώ ότι είναι και τόσο ικανοποιητικό το ποσό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Γιάννη Σκάιερ για αυτό που είπε και για την αναφορά του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Α, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολλά και διαφορετικά μέρη. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στην Αγγλία, αλλά η Ουαλία δεν έχει κάνει πολλά ασφάλματα και αυτό το αναγνωρίζει η Κομισιόν. Ε, αντιθέτως η Ουαλία είναι ο καλός μαθητής για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ε, τώρα, ε, το έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι καλό να μαθαίνει κανείς από τα παθήματα του παρελθόντος. Όντως, ο ε, μέχρι εδώ ο Γκάιερ καλά κάνει και αναφέρει τα λάθη, τα σφάλματα του παρελθόντος, αλλά θα πρέπει να δει λίγο και το μέλλον για το που διατίθεται τα κονδύλια στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο παρακαλώ εσείς. Πείτε το όνομά σα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Γκάιερ, ο οποίο τονίζει δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα τη δυνατότητα διόρθωσης των εποπτικών συστημάτων που προστατεύουν τον προπολογισμό και δεύτερον αναφέρει και την ανάπτυξη μιας νέας νοτροπίας επιδόσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά το πρώτο στοιχείο, την διορθωτική ικανότητα, ξέρετε ότι ο Επίτροπος Έμετα στις 2 Οκτωβρίου θα έρθει στην Επιτροπή σας και θα παρουσιάσει την ανακοίνωσή μας για την προστασία του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Σήμερα βρισκόμαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ανακοίνωσης αυτής και να ξέρετε ότι θα αναφέρει όλα τα σημεία τα οποία εντοπίστηκαν την έκθεση απαλλαγής που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα θα εξηγήσουμε με έναν τρόπο εύκολα κατανοητό, γιατί και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, τις υποχρεώσεις που προβλέπουν δημοσιονομικοί κανονισμοί και οι συνθήκες, αλλά και τομιακοί κανονισμοί, για πρώτα απ' όλα πώς προλαμβάνονται τα σφάλματα και δεύτερον, εφόσον δεν προλαμβάνονται, πώς εντοπίζονται και διορθώνονται. Και εξηγείται εκεί όχι μόνο ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά τι πρέπει να κάνουν και τα κράτη-μέλη. Επίσης θα εξηγήσουμε και την διαδικασία την πολιετή. Τα 4,5 δισεκατομμύρια που αναφέρθηκαν φυσικά έχουν να κάνουν με σφάλματα του παρελθόντος. Το σύστημα όμως θα διασφαλίζει τα σφάλματα τα οποία εντοπίζονται για παράδειγμα για το 2012 θα διορθώνονται στο μέλλον. Δεν θέλω να μπω περισσότερο σε λεπτομέρειες γιατί ο Επίτροπος έμετα ο ίδιος θα σας παρουσιάσει όλες τις λεπτομέρειες της ανακοίνωσης αυτής. Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή την νέα κουλτούρα, τη νέα νοοτροπία επιδόσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όσο αναφέρει η έκθεση Γκάιερ της ε, απαιτήσει που αναφέρονται στη διοργανική συμφωνία για παράδειγμα και θα επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στις εσωτερικές πολιτικές εν ώψη της στρατηγικής 2020 και σε όλους τους τομείς πολιτικής θα συμπεριλάβουμε ενημέρωση ιδιαίτερα στην έκθεσή μας βάσει το άρθρο 318. Ευχαριστούμε πολύ. Με άλλος κανείς θέλει το λόγο παρακαλώ. Ο εισηγητής τότε. Παρακαλώ Γιάννης, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αν θέλουμε να μειώσουμε το, το ποσοστό των σφαλμάτων, των λαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δούμε την κάθε περίπτωση χώρια και να τη μελετήσουμε, να την ελέγξουμε και να προχωρήσουμε στο μέλλον. διαφορετικά, να διορθώσουμε ορισμένα πράγματα. Η ίνγκε έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Κυρίως η περιφερειακή πολιτική είναι αυτή που, στην οποία γίνονται τα περισσότερα σφάλματα έχει δίκιο αλλά γιατί γίνονται τα λάθη αυτά ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι έγινε μία ολόκληρη ιστορία και προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του βασιλείου της Ισπανίας για ποσά τεράστια πολλών ετών. Δεν θα ήταν τώρα δίκαιο να πούμε ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση που έφταιγε για όλα αυτά. Πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά εκείνο που είναι αλήθεια είναι ότι στη Ισπανία αυτή τη σταγμητική αυτή τη στιγμή η σχέση των κεντρικής και των περιφερειακών κυβερνήσεων αν μπορούμε να τις πούμε έτσι ε, η σχέση αυτή δεν είναι και πολύ καλή τι να κάνουμε να πούμε, ζητήσουμε από το Ισπανικό κράτος λοιπόν ε, να φτιάξει τη σχέση του με τις, τη σχέση αυτή μεταξύ κέντρου και περιφερειών. Αυτό θα ήταν πέραν των αρμοδιοτήτων μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή όλη υπόθεση είναι ένα πρόβλημα ε, διαχείρισης ε, το οποίο θα μπορούσε να διορθωθεί με κάποιους πρακτικούς τρόπους ε, και στη Γερμανία, στη Βόρεια Ρινανία, Βεστφαλία, ξέρετε πολύ καλά τι έχει γίνει. Όχι επειδή οι υπάλληλοι της περιφέρειας αυτής είναι ε, διεφθαρμένοι, αλλά γιατί δεν αντιστοιχούν σωστά, δεν συμπίπτουν οι κανόνες που εφαρμόζονται στο κρατήδιο αυτό της Γερμανίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται διόρθωση, χρειάζεται ε, έλεγχος και διόρθωση. Καταλαβαίνετε ότι ε, τα πράγματα είναι περίπλοκα ε, αν θέλουμε πραγματικά να δούμε πού οφείλονται τα σφάλματα, τα λάθη που έγιναν, ε, πρέπει να κάνουμε ακόμη αρκετή δουλειά. Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουμε κάνει ε, ε, μελέτη των επιμέρους σφαλμάτων ένα-ένα, πρέπει να καθίσουμε τώρα με σταυρωμένα τα χέρια και δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Θα ήθελα επίσης να πω γιατί κάποιος ρώτησε το 4,5 δις σε τι χρονική περίοδο αναφέρονται. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς να σας πω, θα σας απαντήσω, αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι να σημειώσετε ότι γίνονται ανακτήσεις και τα ποσά των ανακτήσεων, τώρα χρεωστή τους καταφληθέτων και τα λοιπά συνεχώς αυξάνονται και διορθώνονται με αυτή την έννοια τα λάθη, τα σφάλματα Πρόκειται, η μέθοδος της ανάκτησης είναι μια μέθοδος η οποία λειτουργεί τελικά. Ε. Βεβαίως γίνονται σφάλματα. Λυπηρό αυτό, αλλά η Κομισιόν έχει μηχανισμούς που εκ των υστέρων βοηθούν για να ανακτήσει κάποια ποσά για την κυρία Σεν, Ναι, κοιτάξτε, ο φορολογούμενος πληρώνει στο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος δίνει τα χρήματα στην Κομισιόν και από εκεί και πέρα η Κομισιόν δίνει στα κράτη-μέλη, όχι ένα προς ένα, αλλά μέσω προγραμμάτων κτλ, ε, χρήματα για να προχωρήσουν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ ζητώ και κάποιοι συνάδελφοι μαζί μου το εξής. Αν τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν σωστή διαχείριση η εφαρμογή των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε πρέπει τα προγράμματα αυτά να διακόπτονται, να σταματούν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Ισπανία σταμάτησαν και προγράμματα πέραν των ανακτήσεων. και αν πράγματι αυτά που λέει το Ηνωμένο Βασίλειο σωστά στη γεωργική δαπάνη υπάρχουν, δίνονται ποσά ανεφλόγου πρέπει να ανακτηθούν ή πρέπει να σταματήσουν τα προγράμματα σας υποστηρίζω απόλυτα κυρία Ανδρέσαν Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς θέλει να παρέμβει παρακαλώ Τότε το μόνο που πρέπει να σας πω είναι ότι το κείμενο του Γιάννης Γκάιερ μπορεί ακόμα να τροποποιηθεί. Η προθεσμία είναι η 18 Σεπτεμβρίου για την προθεσμία τροπολογιών. Τετάρτη. Στις 2 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε για την γνωμοδότηση. Καλώς. Καλώς. Οπότε... Πάμε στο τελευταίο σημείο που έχουμε στην ημερήσια διάταξη για σήμερα και είναι η επίσκεψη που θα κάνει αντιπροσωπεία μας 18 με 20 Σεπτεμβρίου στην Βουλγαρία. Η επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Γένς Γκάιερ. Οπότε το λόγο θα δώσω στον Γένς Γκάιερ για να μας πληροφορήσει για την αποστολή αυτή. Για την επίσκεψη αυτή σήμερα προχωρήσαμε γρήγορα Θέλω να πω σε όσους ε, εδώ από την Γραμματεία για το Δικαιό Προσωπικό δεν βλέπουν ε, τους συντονιστές τους στην αίθουσα, ας φροντίσουν να τους ειδοποιήσουν για να μπορέσουμε πιο γρήγορα να αρχίσουμε τη συνεδρίαση των ε, συντονιστών παρακαλώ. Οι σοσιαλιστές, το ΕΛΚ είναι εδώ, οι φιλελεύθεροι επίση, Οι Γκούε, δεν ξέρω, πρέπει να τους βρούμε, ούτε η συντηρητικοί είναι εδώ. Οπότε ας φροντίσουν οι πάλι παρακαλώ να τους βρούνε. Γέννηση για τη Βουλγαρία, πες μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεύτερη επίσκεψη στο Καλίνιγκραντ ε, Πρώτη για μια τότε με τις... Ε, ε, ε, έχουμε πει, είπαμε ότι μας χρειάζεται μια ομάδα η οποία όχι απλώς να θεωρεί γενικώ για την να μιλάει γενικώ θεωρητικά για, τις, ε, ε, για τα ασφάλματα ε, και τα ασφάλματα στην πλευρά των δαπανών. Μετά από εκείνη την επίσκεψη του Καλίνικ λοιπόν, είπαμε ότι όχι λάθος δεν ήταν η δεύτερη επίσκεψη στο Καλίνιγκρα ήταν μετά τις επισκέψεις που έγιναν στην Αμβέρσα και στο Ρότερνταμ που συζητάγαμε το πόσο αποτελεσματικά είναι τα η αποτελεσματική είναι η έλεγχη των εξωτερικών συνόρων με το λαθρεμπόριο κτλ. Ε, τότε λοιπόν είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε και την πλευρά των εσόδων και όχι μόνο των δαπανών τι, τι γίνεται. Ε, και είπαμε ότι θα πρέπει να ελέγξουμε τα εξωτερικά μας σύνορα ε, να δούμε ποιοι είναι οι ευαίσθητοι κρίκοι ποια είναι τα πιο ευάλωτα ποια είναι τα πιο ευάλωτα σύνορα ε, παραδείγματος χάρη που έχουμε πρόβλημα με προϊόντα καπνού ένα δις ε, έσοδα λείπουν ας πούμε από τον καπνό και από το λαθρεμπόριο του, των προϊόντων καπνού ε, δεν πρόκειται για μικρά ποσά πρόκειται για μεγάλα ποσά ε, λοιπόν σιγά, σιγαρέτα και ε, προϊόντα καπνού ε, αυτό ένα μια κατηγορία προϊόντων που υπάρχει τεράστιο λαθρεμπόριο και άλλο, άλλα προϊόντα τα προϊόντα από μίμησης. Ε, και εκεί χάνονται μεγάλα χρήματα και εκεί πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Όπως ξέρετε η Βουλγαρία, η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν σύνορα σε μια περιοχή όπου διαπιστώνεται μεγάλο λαθρεμπόριο ιδιαίτερα προϊόντων καπνού. Είπαμε λοιπόν ότι καλό θα ήταν να οργανώσουμε μία επίσκεψη ε, στην περιοχή για να δούμε ποια είναι η κατάσταση και πού μπορούν να επιτευθούν βελτιώσεις. Φαντάζομαι ότι θα πήρατε το πρόγραμμα βεβαίως πέραν του λαθρεμπορίου εμπορευμάτων και αγαθών γίνεται και λαθρεμπόριο ανθρώπων ε, στα σύνορα αυτά είναι δυστυχές αυτό είναι κρίμα αυτό αλλά συμβαίνει και στο Πάστρο Γκόρ ε, θα ασχοληθούμε θα δούμε το περιφερειακό κέντρο ελέγχου που θα ασχοληθούμε ακριβώς με το θέμα αυτό του, της λαθρέας διακίνησης ανθρώπινων όντων. Είναι ε, <coughs> ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί και ε, η διάσκεψη των Προέδρων και οι ειδικέ κοινοβουλευτικέ επιτροπές ζήτησαν να γίνει η μελέτη αυτή και Βεβαίως αντίστοιχα θα συζητήσουμε και άλλα πράγματα τα οποία θα βρουν, τα πορίσματα για τα οποία θα βρουν το δρόμο τους σε, σε άλλες επιτροπές πέραν της επιτροπής αυτής εδώ. Λοιπόν, είναι μεγάλη η διαδρομή. Ξεκινάμε από τα σύνορα Βουλγαρίας-Τουρκίας, τα σύνορα Βουλγαρίας Ελλάδας δεν είναι μικρή απόσταση ε, πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψη αυτή βεβαίως κρίμα είναι ότι ε, κρίμα είναι που θα τελειώσει η το έργο αυτής, η επίσκεψη αυτή στο, στην Κωνσταντινούπολη στο τέλος της, ε, ε, του ταξιδιού μας ε, θα γίνει η συνέντευξη τύπου εκεί στο Ισταμπούλ ε, ίσως θα πρέπει να επαναλάβουμε ορισμένα πράγματα όταν γυρίσουμε εδώ ίσως θα πρέπει να παρουσιάσουμε από κοινού τα αποτελέσματα αυτού του ταξιδιού με αυτά του ταξιδιού στο Καλίνιγκρατ. Ευχα, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κανένα συνάδελφος μήπως που θέλει κάτι να πει. Παρακαλώ. Και εκπρόσωποι της Όλαφ ε, είναι αν θέλετε κάτι. Παρακαλώ κύριε Μιλντορφ. Ευχαριστώ. Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένω αυτήν την αποστολή. Θυμάμαι ότι μετά από την ε, παρόμοια ε, αποστολή στο Καλίνιγκραντ ζητήσαμε μέσω προφορικής ερώτησης από το... και μέσω του Προεδρείου να κάνει η Κομισιόν και το Συμβούλιο ε, ανακοίνωση σχετικά με το λαθρεμπόριο τσιγάρων ε, από το Καλίνιγκραντ. Νομίζω ότι ε, πρέπει να δούμε τι έγινε με αυτήν την, το ερώτημα προς διάσκεψη των Προέδρων. Προωθήθηκε το ερώτημα αυτό. Η κυρία Γκρέσλερ, θα το συζητήσω με τη γραμματεία και θα δούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσοι οι διερμηνείς θα είναι μαζί. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εμείς σαν επιμέρους, σαν μέλη της ομάδας αυτής ε, δεν πρέπει να πάρουμε διερμηνείς ο καθένας. Δεν πρέπει να είναι χιλιάδες οι διερμηνείς εκεί. για το λαθρεμπόριο σιγαρέτων, από ό,τι φαίνεται ακόμα δεν έχει προχωρήσει, θα το συζητήσουμε στους συντονιστές. Τώρα, η Επιτροπή, μου είπε ο κύριος Ντόμπο από τη Γενική Διεύθυνση Home, ο κύριος Κατάνια και Σόντος από την Όλαφ επίσης. Κάποιος από αυτούς, η περισσότεροι, παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Ε, είμαι από την DigiHome. Είμαι από την ε, DigiHome. Είμαι από την DigiHome. Καλωσορίζει η Κομισιόν αυτήν την επίσκεψη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ε, στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας-Βουλγαρίας. Να πιστήσω την προσοχή σας ότι αυτά τα χερσαία σύνορα είναι ε, ε, σύνορα τα οποία παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα όσον αφορά την λαθρομετανάστευση, κυρίως και λόγω της καταστάσεως στην Συρία. Έχουμε λοιπόν αυξημένο κύμα μεταναστών και τούντων άσυλο από την Συρία. Η υπηρεσία Frontex, να σας πω, ότι συντονίζει την λεγόμενη κοινή ε, επιχείρηση μαζί με τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, την λεγόμενη χερσαία επιχείρηση Ποσειδών ε, ε, Ξηράς. Ε, βεβαίως υπάρχουν και άλλες έκνομες πράξεις οι οποίες συνδέονται με το πέρασμα των συνόρων, αυτών των εξωτερικών συνόρων όπως ας πούμε λαθρεμπόριο σιγαρέτων και άλλων. Ε, πάντως θα είναι και μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε να γίνει και συζήτηση όσον αφορά την διαχείριση των χερσαίων συνόρων ε, της Βουλγαρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ενδιαφέρον. Όλαφ, θέλετε κι εσείς να παρέμβετε παρακαλώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλό απόγευμα, Σαλβατόρε Κατάνια από την Όλαφ. Επικεφαλής των παρα... του παραχαραγμένων προϊόντων και προϊόντων καπνού. τα χερσαία σύνορα και η οδική γραμμή διασύνδεση ε, στο σημείο αυτό δεν είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο. Από την Αμόχωστο όμως ε, μέχρι τα θαλάσσια σύνορα έχουμε πρόβλημα ε, με την... με την το λαθρεμπόριο μέσω θαλάσσης. Έχουμε ε, μεγάλη ανταλλαγή πληροφοριών ε, με την Τουρκία όσον αφορά τα εμπορικά ε, πλοία τα οποία ακολουθούν αυτήν την ακτογραμμή. Ένα δις παράνομα τσιγάρα έχουν μπει το πρώτο εξάμεινο του 2013 από την Αμόχωστο, το ελεύθερο λιμάνι της Αμόχωστου ε, προς την ε, Ευρώπη. Ε, είχαμε κατάσχεση δύο σκαφών που ξεκίνησαν από την Αμόχωστο. Ε, κατάσχεση η οποία έγινε από τις ε, τουρκικές αρχές που βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν την κατάσχεση λόγω της μεταφόρτωσης σε ανοιχτή θάλασσα από το ένα πλοίο στο άλλο του παράνομου φορτίου. Ε, στο δεύτερο εξάμεινο είχαμε μονάχα ε, ένα φορτίο 10 εκατομμυρίων σιγαρέτων που ξεκίνησε από την ε, αμόχωστο. Επίσης, επανερχόμενος σε τα χερσαία οδικά σύνορα είναι πολύ ε, μικρά πρέπει να πω στην έκταση και όσον αφορά ε, την ε, παράνομη διακίνηση σιγαρέτων για μας ευαίσθητο σημείο είναι ο λιμένας του Μπουργκάς. Ε, πρόκειται για φορτία τα οποία φορτώνονται κυρίως στο port site της Αιγύπτου ε, και θα έπρεπε να φτάσουν στο Μπούργας αλλά τελικά δεν έφτασαν ποτέ ε, πράγμα που σημαίνει ότι άλλαξαν πορεία μεσοπέλαγα και επομένως ήταν λάθος τα στοιχεία φόρτωσης όσον αφορά τις κατασχέσεις ε, σιγαρέτων και όσον αφορά ε, την ε, κατάταξη αναμέγεθος και αναποσό κατάσχεσης. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τη Βουλγαρία. Μας δίνουν πάντοτε λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά την, τις πληροφορίες για τις έκνομες δραστηριότητες και τις εγκληματικές ομάδες. Επίσης έχουμε έχουμε και διάφορους, ε, διάφορες εγκληματικές οργανώσεις ε, οι οποίες ε, κυκλικά, ομόκεντρα μάλλον δουλεύουν με τη Βουλγαρία και κυρίως με την Αλβανία. Πρέπει να σας πω ότι και με την Τουρκία έχουμε εξαιρετική συνεργασία, άλλωστε ανέφερα και προηγουμένως τις περιπτώσεις κατάσχεσης σιγαρέτων που ξεκίνησαν από την αμόχωστο και έγιναν από τις τουρκικές αρχές. Επίσης, δύο λόγια για την κατάσταση των ε, σκαφών ε, και τις πληροφορίες τις οποίες ε, παίρνουμε σε στενή συνεργασία με τους ε, με τις χώρες να αναφέρω την υπόθεση του σκάφους Άνταμ, γνωστό για την φόρτωση παρανόμων σιγαρέτων από την ε, Αμόχος. Το Χάθηκε ε, για ένα, χρο... για ένα μήνα συγγνώμη, αυτό το πλοίο μέχρι ότου τον Απρίλιο του 2013 η Guardia di Finanza της Ιταλίας το ε, ε, βρήκε στην Παντελερία, στα στενά της ε, Παντελερίας, φορτωμένο με πολλά παράνομα σιγαρέτα, καθώς επίσης και ναρκωτικές ουσίες. Αυτά ήθελα να σας πω και βεβαίως μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Κατάνια. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Είναι καλό να έχουμε όλες αυτές τις προφορίες για την αντιπροσωπεία μας. Αν αυτά που μας είπατε μπορείτε να μας τα δώσετε και γραπτά, τα speaking notes δηλαδή που είχατε, θα μπορούσαμε να τα επισυνάψουμε στο πρόγραμμα, να τα πάρουν οι ευρωβουλευτές, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους ευρωβουλευτές. Ο Ντι Κρέσλερ και ο κύριος Γκάιερ είναι επόμενο μιλητή. Παρακαλώ κύριο Ντί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό οι ευρωβουλευτές να μπορούν και να πηγαίνουν να ελέγχουν από κοντά πόσο καλά λειτουργούν τα εξωτερικά μας σύνορα. Γιατί οι πολίτες θεωρούν ότι είναι μία από τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελωνία λοιπόν που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις συνθήκες έχουν έναν τρόπο λειτουργίας όπου είναι οι εθνικές αρχές που κάνουν τη δουλειά των τελωνίων και στέλνουν το λογαριασμό μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να πάμε και να δούμε από πρώτο χέρι την ποιότητα της δουλειάς που κάνουν ε, οι τελωνιακοί επιτόπου. Στην προηγούμενη θητεία από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ετοιμάσαμε έκθεση για ένα τελωνιακό σύστημα που διαπιστώναμε πως δεν ήταν ικανοποιητικής ποιότητας. Και είχα προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μία πρόταση για να εξευρωπαϊστούν τα τελωνία. Με την έννοια να μην είναι υπό τις κυβερνήσεις των χωρών μελών, αλλά υπό τις ευρωπαϊκές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν νομίζω να έκανε ποτέ μια τέτοια μελέτη. Κρίμα. Υπό το φως πάντως των όσων θα διαπιστώσετε επιτόπου και εφόσον συμφωνήσουν οι πολιτικές ομάδες, ίσως καλό θα ήταν να επανέλθουμε σε αυτή την ιδέα. Και επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε γι' αυτό να είμαστε αποτελεσματικοί αλλά η αποτελεσματική θα εξαρτηθεί από μία αρχή που θα είναι επικεφαλής και όχι πολλών. Ευχαριστούμε κύριε Γκρέσλερ. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Κατάνια, έχω αρχίσει να αμφισβητώ κατά πόσον ε, αυτή τα, τα κοινά σύνορα ε, και η σχετική η ιδέα αυτών των ανοιχτών αν θέλετε συνόρων είναι καλή όχι γιατί το, δεν ξέρω αν το θυμάστε και από την επίσκεψη του Καλίνιγκραντ κουβεντιάζαμε ακριβώ για τα σύνορα με την Μολονία και τα λοιπά. Λοιπόν, ερώτηση προς τον κύριο Κατάνια. Κατάσχεση ενός εκατομμυρίου σιγαρέτων έγινε μέχρι τώρα. Τι ήτανε συγκεκριμένα τσιγάρα, συγκεκριμένες μάρκες τσιγάρων ή ήταν λαθρέα τσιγάρα που, με άσχετες μάρκες. Πρόκειται για μάρκες που τις πληρώνει, δηλαδή τις αγοράζει ο Ευρωπαίος πολίτης ή όχι. Ε, Επίσης η Βουλγαρία δεν είναι μόνο, δεν εισάγει μόνο λαθρέα προϊόντα αν θέλετε είναι και χώρα διαμετακόμισης, transit και τι ρόλο παίζουν θαλάσσιες μεταφορές, τι ρόλο παίζουν χερσαίες μεταφορές. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις από την κυρία Γκρέσλερ. Έχετε ο κύριος Γκάιερ να ρωτήσει ρωτήσω μια παραλλαγή είναι η ερώτησή μου των ερωτήσεων της Ίγκε αν θυμάμαι καλά η, αν η επιλογή των ε, θεμάτων αν θέλετε και των τόπων επίσκεψης της ομάδας μας έγινε με βάση κάποια στοιχεία από την Ευρωπόλη η οποία Ευρωπόλ κάθισε και είδε ποιοι είναι οι συνήθεις δρόμοι του λαθρεμπορίου για ορισμένα προϊόντα κτλ. Ένα θύλακας ήταν το Καλίνιγκραντ, μια άλλη περιοχή είναι αυτή που θα επισκεφθούμε τώρα. Ο Κατάνια λέει ότι παίζει ρόλο και, το, ε, και οι δαλάσσιες μεταφορές ε, Κύπρο ε, Τουρκία και τα λοιπά. Ναι, άρα τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά όπως τα παρουσίασε η Ευρωπόλ. Ρωτώ λοιπόν, τα στοιχεία που μας δώσατε είναι μόνο για προϊόντα καπνού, για λαθρεμπόρια προϊόντων καπνού, είναι γενικώ για προϊόντα, για εμπορεύματα και για το εμπόριο ανθρώπων ας πούμε πρόκειται για λαθρομετανάστευση για λαθρομετανάστες που τους ε, συλλαμβάνουμε στα σύνορα ή, περί τίνος ακριβώς πρόκειται Τρεις ερωτήσεις λοιπόν, δυο από την κυρία Γκράσσερ μία από τον Γκάιερ. Μπορεί να απαντήσει ο κύριος Κατάνια. Παρακαλώ. Thank you, Mr. <clears throat> Concerning Bulgaria. Ε, Όσον αφορά την ε, Βουλγαρία, Πρόκειται για χώρα διαμετακόμισης αλλά και χώρα ε, ε, εκκίνησης φορτίων ε, σιγαρέτων. Όσον αφορά τις μάρκες, πρέπει να σας πω ότι μπορώ να σας πω αργότερα ποιες είναι οι πιο κατασχεμένες ε, ε, μάρκες ε, τσιγάρων. Από την άλλη πλευρά βέβαια μπορούμε να βρούμε και τις μάρκες τις οποίες περισσότερο ζητούν οι χώρες προορισμού όσον αφορά τις θαλάσσιες οδούς για το λαθρεμπόριο σιγαρέτων. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μεγάλα ποσοστά αυτών των σιγαρέτων μεταφέρονται ε, ε, ε, με, πλοία. Έχουμε 22 κατασχέσεις 22 εκατομμυρίων μεγάλων κουτιών, master boxes σιγαρέτων. Επίσης, 25 27 συγγνώμη, φορτία έχουν κατασχεθεί στην Ελλάδα. Ε, επίσης ε, έχουμε παλιά πλοία ε, τα οποία έχουν σημαίες του Μπελίς, του Παναμά ή άλλων περιέργων νήσων, πλοία τα οποία ξεκινούν από το Μπουργκάς και που ε, βρίσκονται στη θάλασσα για μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθώντας να βρουν ένα άνοιγμα ε, για να ξεφορτώσουν το φορτίο τους. 20 ε, λεπτά χρειάζονται σε ένα μικρό λιμάνι στην Ιταλία, στην Ισπανία ή στην Ελλάδα για να ανοίξουν τον καταπέλτη και να ξεφορτώσουν το, το φορτίο. 20 λεπτά οχτώ ε, φορτηγά τα οποία ήταν γεμάτα ε, ε, με, με, με τέτοιου είδους προϊόντα φορτωμένα σε ένα φέρι 20 λεπτά κάνανε να τα φορτώσουν, να τα ξεφορτώσουν και να γεμίσουν 8 φορτία. Επίσης και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουμε ε, παράνομα ε, εργαστήρια ε, και πρέπει να σας πω ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση στην Λιβύη είχαμε αυτόματα αύξηση της εκκίνησης ε, ε, τσιγάρων παρανόμων προς την ε, Λιβύη. Εκατοντάδες χιλιάδες τσιγάρα παράνομα μεταφέρονται στη Λιβύη, όμως δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, αν, έχουν, αν κατασκευάζονται εκεί. Ένας άλλος προορισμός είναι η Τινησία. Είχαμε ε, πέντε κοντέινερ από το Port Said προς ε, την, Ισία. Οι συνάδελφοι των ε, την τελωνίων ε, ανέφεραν ότι ουδέποτε αυτά τα πλοία, αυτό το φορτίο μάλλον δεν έφτασε ε, εις την, ε, Προφανώς λοιπόν έγινε μεταφόρτωση στα ανοιχτά. Πολλά είναι επίσης τα σκάφη τα οποία φεύγουν από τον πατούμι της ε, Γεωργίας, ε, καταπλέουν, ε, μάλλον διαπλέουν την Μαύρη Θάλασσα, γιατί και εκεί έχουμε τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που βλέπουν την Μαύρη Θάλασσα που είναι ευαίσθητη ζώνη. Να σας πω τα εξής επίσης. Ε, πολύ πρόσφατα είχαμε την πρώτη κατάσχεση, ε, κατάσχεση ε, ενός μιας ενός ταχύπλοου από το Μαυροβούνιο μέχρι το 2000 από την περίφημη υπόθεση λαθρεμπορίας σιγαρέτων από το Μοντενέγρο στην Ιταλία δεν είχαμε ξανακάνει τέτοιου είδους μεγάλη κατάσχεση. Ε, ελπίζω ότι δεν θα ξαναρχίσουμε ένα καινούριο κύμα φόρτωσης ταχυπλών από το Μαυροβούνιο με ε, κατεύθυνση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να σας δώσω και κάποια αριθμητικά στοιχεία για την τρίτη ερώτηση. Οι Αφρικές, ε, ε, στις αφρικανικές χώρες ε, έχουμε τεράστιες ποσότητες διακινούμενων σιγαρέτων. Από την στη Μαυριτανία, ας πούμε, από την Πάλμας, είχαμε πληροφορίες για την φόρτωση 20 containers προς την Μαυριτανία. Προφανώς ε, πρόκειται για premium τσιγάρα καλής ποιότητα και προφανώς ε, δεν αφορούσαν ε, την εσωτερική αγορά της Μαυριτανίας. Μέσω της Σαχάρας προφανώς θα ξαναπεράσουν από τη Βόρεια Αφρική για να βρουν το δρόμο τους να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συρία επίσης στο παρελθόν ήταν χώρα διαμετακόμισης τώρα. Έχουν κλείσει τα σύνορα λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχει εισάγει η Συρία από το 2011, 27 ε, Μαΐου και εποπλέον αναγκάστηκαν ε, και οι λαθρέμποροι να αλλάξουν διαδρομές. Για να απαντήσω συνολικά στην τρίτη ερώτηση μπορώ να σας πω κάποια στατιστικά στοιχεία. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι συλλέγουμε στατιστικές από τα κράτη-μέλη τα οποία μας δίνουν πληροφορίες όσον αφορά τις ε, κατασχέσεις ε, κάθε τρεις ε, μήνες. Αλλά οι κατασχέσεις αναφέρονται μονάχα σε προϊόντα καπνού, συγκεκριμένα δεν σε σιγαρέτα. Είτε πρόκειται για κανονικά τσιγάρα, είτε για παραχαραγμένα. Παράδειγμα, το 2012 στη Βουλγαρία οι κατασχέσεις ήταν περίπου της τάξεως των 83 εκατομμυρίων σιγαρέτων. Και βεβαίως εμείς δίνουμε όλα τα στοιχεία αυτά, κάνοντας και κάποιες κατατάξεις ε, όχι μόνο βάσει των κατασκευμένων ποσοτήτων αλλά και βάσει των ε, ε, μαρκών των τσιγάρων. Καθώς επίσης και βάσει των στοιχείων που έχουμε όσον αφορά τους χώρε τις χώρες προορισμού. Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις. Κυρία Γκρέσλερ. Είδατε λοιπόν κυρία Κατάνια το κακό ε, βασιλεύει. Εδώ όμως θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη Βουλγαρία. Ρωτώ, τι ρόλο παίζει η Βουλγαρία εδώ. Τι μας λέτε, ε, δεύτερη θέση στο λαθρεμπόριο. Τι να σας πω. Ρωτώ, ποια είναι αυτά τα τσιγάρα, τι τσιγάρα είναι αυτά που κυκλοφορούν στη Βουλγαρία, θα θέλαμε μια απάντηση, όχι τώρα βέβαια, αλλά κάποια στιγμή να μας δώσετε γρήγορα τα στοιχεία. Μετά αναφερθήκατε στη Συρία, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκίνησε η Όλαφ μια υπόθεση εδώ πριν από καιρό για τη Συρία. Ερώτηση, επειδή έχει περάσει κάμποσος καιρός, ε, τι έγινε με αυτή την υπόθεση στη Συρία και άλλο ερώτημα πόσες υποθέσεις πραγματεύεται ο Όλαφ όσον αφορά λαθρεμπόριο τσιγάρων. Η τελευταία είναι ενδιαφέρουσα βέβαια ερώτηση αυτή για τη Συρία. Υπάρχει και γραπτή ερώτηση. Κύριε Κατάνια, για την τελευταία αυτή ερώτηση της κυρίας Γκρέσλ, μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ. Eh, eh, ε, πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά την ε, Βουλγαρία ε, η υποθέσεις βρίσκονται υπό ε, έλεγχο. Όσον αφορά την Συρία, ε, έχουν αναφερθεί παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων ε, που έχει εφαρμόσει η Συρία. Επίσης και στην Κύπρο σε στενή συνεργασία με τις κυβερνητικές κυπριακές τελωνιακές αρχές, σε συνεργασία με την Όλαφ βέβαια, έχουν καταγραφεί απόπλη πλοίων μετά από την εγκαθίδρυση αυτών των περιοριστικών μέτρων όσον να σας πω επίσης ότι η Όλαφ δεν είναι αρμόδια για την ε, διερεύνηση ε, της, ε, των περιπτώσεων παραβίασης των περιοριστικών μέτρων προς την Σύρια. Απλώς εμείς ζητούμε σε περίπτωση καταγραφής τέτοιων περιστατικών να υπάρχει η ενημέρωση της μόνιμης αντιπροσωπείας της Κύπρου περί αυτού. Επίσης όσον αφορά τις μάρκες των κατασχεθέντων προϊόντων, δεν τις έχω εδώ, ε, αλλά θα σας δώσω το συντομότερο δυνατόν τα στοιχεία αυτά, γιατί πρέπει να σας πω ότι τα κράτη-μέλη μας δίνουν όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή όσον αφορά τις μάρκες των κατασχεμένων τσιγάρων. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε πληροφορίες, ε, έχουμε πάντα πληροφορίες για τον αριθμό των κατασχέσεων, αλλά όχι πάντα και από όλες τις χώρες μέλη ε, για τη μάρκα των ε, κατασχεμένων ε, τσιγάρων. Επομένως, να πω για μία ακόμα φορά ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που μας δίνουν τα στοιχεία. Εξαρτώμεθα από τα στοιχεία που μας δίνουν. Καλώ άλλε ερωτήσει. Όχι? Κύριε Γκάι, τίποτα. Μπορούμε να τελειώσουμε, να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Ωραία, δεν υπήρξε απάντηση. Αλλά ο κύριο Κατάνια, δίχω άλλο, θα φροντίσει και ίσως τις speaking notes του το γραπτό σημείωμα που μας παρουσίασε σήμερα θα συμπεριλάβει ίσως και κάτι σχετικά με την ερώτηση αυτή. Αυτά έτσι ολοκληρώθηκε η μερική διάταξη για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους. Αύριο στις 9 θα αρχίσουμε. Τώρα συνεδρίαση συντονιστών και κλεισμένο το θυρών, έτσι. Άντε 10 λεπτά διάλειμμα και στις 5 παρα 10 θα αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών.